habe zwei Änderungen Αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη αναβάλλεται η έκθεση Καβαντά για τον Ιούλιο. Ούτω ή άλλω έχουμε μικρό χρονικό διάστημα για αυτή την αναβολή και δεν είναι και τόσο κατεπήγον. Παρακαλώ, συνάδελφοι που ασχολείστε με αυτό, να συνεργαστείτε επικοδομητικά. Δεύτερον, κατά την αρχή τη ημερήσια διάταξη, σήμερα το απόγευμα θα ήθελα ένα σύντομο σημείο να μπορέσει να ενταχθεί για την Europe for Citizens στην Ευρώπη για τους πολίτες, ώστε την παρουσία της Επιτρόπου Βασιλείου το απόγευμα να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τι αποφάσισαν οι συντονιστές για την Ευρώπη για τους πολίτες και τι θα κάνουμε για το Europe for Citizens και τι έχουμε αποφασίσει σχετικά. Για αυτή την ημερήσια, αλλαγή της ημερήσια διάταξης υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Τα πρακτικά της τελευταίας μας συνεδρίασης θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται αν δεν υπάρχουν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης κάποιες ενστάσεις ή αλλαγές. Στο σημείο 3 σήμερα βρισκόμαστε σε μικρή αίθουσα με λίγες δυνατότητες διερμηνίας και γι' αυτό δεν έχουμε ούτε βουλγαρικά, ούτε τσέχικα, ούτε εσθονικά, ούτε λιθουανικά, ούτε μαλτέζικα, πορτογαλικά και σλοβένικα. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμες. Ολλανδικά μπορείτε να μιλήσετε, αλλά δεν θα υπάρχει διερμηνία προς τα Ολλανδικά. Ζητώ συγγνώμη για τους συναδέλφους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γλώσσες τους ε, αλλά η Ματούλα νομίζω, Ματούλα αφοράται μόνο και οι άλλοι μπορούν να μιλήσουν στην ε, γλώσσα τους. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4. Το 4 αναβλήθηκε όπως είπα, εντάξει. Και κανένας από εσά δεν εξέφρασε κάποια ένσταση. Όλοι συμφωνήσατε. Περνάμε στο 5 και 6 τώρα. Αυτά τα δύο σημεία θα τα εξετάσουμε από κοινού το 5 και το 6. Είναι τα σημεία που αφορούν τα διαθωτικά ταμεία αυτά τα δύο θέματα και η συγκήτριά μας είναι η κυρία Μπέναραμπ Ατού και στην προηγούμενη συνεδρίαση εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά. Και όλοι είχαμε ευκαιρία να καταθέσουμε τροπολογίες όσοι επιθυμούσαμε. 50 τέτοιες τροπολογίες κατατέθηκαν για την κοινή θέση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και 70 τροπολογίες ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρωτού ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Μπεναράμπα του. Έχετε τον λόγο κυρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα Απλά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ε, όλους όσους ε, συνεργάστηκαν μαζί μου με τρόπο επικοδομητικό και ευχάριστο για την υποβολή των τροπολογιών και να ευχαριστήσω και την κυρία Φαμπία Φοντανέλη η οποία συνεργάστηκε εξαιρετικά μαζί μας. Κάναμε από κοινού την εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πενεναπατού η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αναφερθεί στο θέμα τον Ιούλιο και ελπίζουμε οι δικέ μα παρατηρήσει να ληφθούν υπόψη. Αυτέ που θα εγκρίνουμε τώρα στην ψηφοφορία, να ενταχθούν στην έκθεση. Περνάμε και ψηφίζουμε. Ελπίζω ότι έχετε όλοι και όλε τι κάρτε σα. Καμιά φορά δεν ξέρει κανεί τι συμβαίνει. Συμβιβασμό 1. Όχι, δεν είναι αυτό. Μια στιγμή. ράμπα του. Πού είναι αυτό εδώ. Ωραία. Συγγνώμη σα ζητώ. Τροπολογία. Δύο καταλόγου έχουμε, είπατε. το πρώτο να πάρουμε. Μάλιστα, πολύ καλά, το βρήκαμε. Άρθρο 2, παράγραφος 2. Είναι αυτός ο κατάλογος, voting list. Τον έχετε αυτόν τον κατάλογο ψηφοφορίας. Εντάξει, όλα εντάξει. Ξεκινάμε με το άρθρο 2, παράγραφο 2, τροπολογία 40, υπέρ τη 40. Όχι, όχι, σε δύο τμήματα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό 2. Μάλιστα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 10. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα. Όμως η Σαμπίνε δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι αφού δεν ψήφισε. Ε, αρχίζει πάλι η ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 10-10 ισοψηφία απορρίφθηκε. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 46 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 48, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ 2 εναντίον. Εγκρίθηκε έτσι. Μάλιστα. Δεν σηκώσατε τα χέρια σας, αλλά είναι νωρίς. Μπορείτε να κάνετε νωρίς ε, τη γυμναστική σας. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 49 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 51 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 51 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 10 υπέρ 12 εναντίον απορρίφθηκε 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 54 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 αποσύρθηκε 57 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 57. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 10 υπέρ 13 εναντίον. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Α, καταπίπτει λέτε. Ωραία, καταπίπτει. Πολύ καλά, συγγνώμη. 58 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην 63 τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Φοπολογία 1 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμό 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 τροπολογία, 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τι είπατε? Να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 32. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 22 εναντίον, κανείς υπέρ. Απορρίφθηκε. Μάλιστα, είναι αστείο πραγματικά, τι να κάνουμε. Α, αυτά, είναι τα γυαλιά που δεν φορούσατε ίσως, τι να πω, εντάξει, γι' αυτό δεν το είδατε. Καταπίπτει η επόμενη τροπολογία και πάμε στην 31. 31 υπέρ, κατά, όχι. Και πάλι. 31 σε δύο τμήματα. Σε δύο τμήματα μάλιστα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 33 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μάλιστα, νομίζω τελειώσαμε έτσι. Τελική ψηφοφορία τώρα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 21 υπέρ, κανείς εναντίον, δύο αποχές. Ευχαριστούμε κυρία Μπένα Ραμπατού. Δουλέψατε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε. Περνάμε στο δεύτερο κείμενο Μπένα Ραμπατού. Αρχίσει με την τροπολογία 22 η ψηφοφορία. Έχετε όλοι έτσι τον κατάλογο ψηφοφορίας. 22 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Λυπούμε Λότα Μπίσκι για τις αποτυχίες. 25 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα. 24 υπέρ, κανείς εναντίον. Δεν φταίω εγώ. Όταν είπα κατά, ο Μάρκο καταψήφισε. Ίσως όμως έφταιγε το ότι μίλησα πολύ γρήγορα. Τι να πω, εγκρίθηκε κανείς εναντίον. Εξαιρετικά. 26 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 30. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Της Καταλήν Σορίν Ιβαν. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 11 υπέρ 13 εναντίον απορρίφθηκε. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 34 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 35 υπέρ κατά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 35 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ 12 εναντίον. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 37 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 39 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Λότα Μπίσκι τι έχουν εναντίον σας. Οι έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την έξι. Ψηφίζουμε την έξι. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 13 εναντίον 12 υπέρ απορρίφθηκε. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 8. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ 11 εναντίον εγκρίθηκε. Θα πάρουμε την 9 τώρα, τι κάνουμε. Η 8 ήταν. Περνάμε στην 9 τώρα. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 49 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 11 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 11 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 14 υπέρ 11 εναντίον εγκρίθηκε 12 υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία εγκρίθηκε 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 13 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 13 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 13 υπέρ 11 εναντίον εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 18 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία, άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 25 υπέρ, κανείς εναντίον, δύο αποχές. Εγκρίθηκε. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Μπένα Ραμπατού. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει αυτό να περάσει και να ληφθεί υπόψη όταν τον Ιούλιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα γίνει η ψηφοφορία εκεί. Και έτσι περνάμε τώρα στο 7. Κυρία Πρόεδρε, να πω δύο λόγια. Θα ήθελα να επιμείνω στο εξή. Ψηφίσαμε για την γνωμοδότηση την έκθεση FSE που αφορά κυρίως την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ε, και επίσης ε, θα κάνουμε και την γνωμοδότηση για τα διορθωτικά ταμεία για την Επιτροπή για την Επιτροπή Ρέτζι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποβάλουμε γνωμοδοτήσεις ε, στην Επιτροπή μας, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ε, μας βλέπουν λίγο σαν διακοσμητική Επιτροπή, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε σημαντική και σωστή χρηματοδότηση οι οποίες θα στηρίξουν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή τις κοινωνικές υποθέσεις. Και εμείς από πλευράς μας έχουμε κάτι πολύ σοβαρό να πούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, τους συναδέλφους σας στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων να τους επιστήσετε την προσοχή ότι οι τροπολογίες μας είναι σημαντικές και πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εγκριθούν. Διότι όπως έχουν τα πράγματα τώρα τα διαρθρωτικά ταμεία δεν είναι έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά σε όλες τις πτυχές. Χρειαζόμαστε για αντιστάθμιση για εκείνα που δεν έχουμε στο πρόγραμμα κατάρτισης για την επαγγελματική κατάρτιση. Πολλά θέματα απεμπολίσαμε και, μας, και είπαμε ότι πρέπει αυτά στο κοινωνικό ταμείο να καλυφθούν και να ενταχθούν. Πρέπει να δούμε, θα ενταχθούν ή όχι. Έχουμε τροπολογίες γι' αυτό. Το άλλο θέμα, το θέμα πολιτισμού, ούτε και αυτό ρητά de facto είχε συμπεριληφθεί. Και ξέρουμε για τις πολιτισμικές δυνατότητες για αυτά τα προγράμματα πολλά μπόρεσαν και μπορούν να επιτευχθούν. Για την Πολωνία έτσι τυχαία ας λάβουμε υπόψη. Και για τους κινηματογράφους στην, Ήπεθρο πληρώθηκαν πρωτοβουλίες και έτσι αυτός ο χώρος της Ήπεθρου δεν αποψηλώθηκε. Διότι οι νέοι έμειναν, παρέμειναν εκεί. Γιατί είχαν κάτι και το βράδυ, ένα κινηματογράφο να πάνε να δουν ένα έργο. Και έτσι αυτό είναι θετικό. Ένα μικρό παράδειγμα είναι αυτό, αλλά πολλά άλλα θα μπορούσα να παριθμίσω. Όπου το, το θέμα του πολιτισμική πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις διαρθρωτικές μεταβολές. Ευχαριστώ την κυρία κυρία Μπεναραμπατού που τα κατάφερε και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους στις κοινοβουλευτικές σας ομάδες να δώσετε μάχη οι απόψεις μας να αντανακλώνται στα ουσιαστικά προγράμματα που θα εγκριθούν. Και πάλι σας ευχαριστούμε κυρία Μπεναραμπατού. Περνάμε τώρα στο μέσο γειτονίας. Ο εισηγητής είναι ο Ιωσήφ Ματουλά. Ο κύριος Μάτουλα την έκθεσή του ήδη μας την έχει ε, καταθέσει τον Απρίλιο και έχουμε τροπολογίες που κατατέθηκαν, 32 συνολικά τον αριθμό. Ο κύριε Μάτουλα, θέλετε να λάβετε τον λόγο να παρέμβετε ή να ψηφίσουμε κατευθείαν. Τι λέτε. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν αμέσως στην έκθεση του Ιωσήφ Μάτουλα. <laughs> Ξεκινάμε. Τροπολογία 23, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 24, υπέρ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 αποχές εγκρίθηκε. 36 υπέρ κατά αποχές αποχές εγκρίθηκε. 37 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 37. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ 11, 11 εναντίον εγκρίθηκε. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Όχι. Α, και πάλι λοιπόν θα ελέγξουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη δεν πρόσεχα. Θα ψηφίσουμε ξανά την 5. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά αυτή τη φορά. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ 12 εναντίον εγκρίθηκε. 6 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 9 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 9 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 15 υπέρ 11 εναντίον εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 11 υπέρ όχι λάθος λέει αν, εγκρι... αν εγκριθεί πάμε στη 12. Εγκρίθηκε λοιπόν αυτή. Α, όχι, δεν εγκρίθηκε. Καταψηφίστηκε, συγγνώμη. 12 λοιπόν, υπέρ. Μόλις το είπα πριν, να πάμε στη 12. 11 είπατε, 11 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 12, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 1 με προφορική τροποποίηση του εισηγητή είναι κάποιος εναντίον όχι λοιπόν υπέρ της 1 δι, ε, κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τροπολογία 1 αυτήν ψηφίζουμε Πέρας ψηφοφορία, 18 υπέρ, 7 εναντίον εγκρίθηκε. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε τώρα ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 18-7 εγκρίθηκε και πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία αυτή πέρας ψηφοφορίας Αποτέλεσμα 25 υπέρ, κανεί εναντίον, μία αποχή. Εγκρίθηκε λοιπόν. Σα ευχαριστούμε πολύ. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Μάτουλα. Και περνάμε τώρα στο σημείο 8 τη ημερησία διάταξη. Περί τίνος πρόκειται εδώ <clears throat> για τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότυπες διευθετήσεις έχει τον λόγο ο κύριος Μιγκάλσκι. Παρακαλώ κύριε Μιγκάλσκι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 na linię, na linię medium, którego jest właścicielem. Zgłaszam taką poprawkę ustną. Παρακαλώ, Ιβο, εσείς έχετε τον λόγο. Respect for the rapporteur and with all sympathy, sympathy but we feel obliged. Αισθανόμαι την υποχρέωση να είμαι να εκφράσω την αντίθεσή μου στην προφορική τροπολογία. Συμβαίνει το εξή. Αν υπάρχει μια ένσταση, η προφορική τροπολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Είμαι σίγουρη όμω, κύριε Μιγκάσκη, ότι ακόμα κι αν είχε γίνει δεκτή αυτή η προφορική τροποποίηση, θα είχε καταψηφιστεί. Πιστεύω ότι η ελευθερία των, των δημοσιογράφων δεν μπορεί να αμφισβητείται από του ιδιοκτήτε των μέσων. Αυτό απλά και μόνο έτσι ω προστίκη. Λοιπόν, τροπολογία 61 αποσύρθηκε. Εντάξει, ψηφίζουμε με 72 πόσες είναι τροπολογίες, 74 τροπολογίες. Εντάξει, συμβιβασμός 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Επτά δεν είναι. Ποιο είναι. Τρία τώρα. Τρία έτσι. Ωραία. Συμβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 14 τώρα. Τροπολογία 14 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε 16 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 10 εναντίον εγκρίθηκε. 19 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 22 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 46 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Αποτέλεσμα 21 υπέρ 6 εναντίον εγκρίθηκε. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 48 και 49. Όχι, ναι, είναι ταυτόσιμες και οι δύο. Υπέρ τη 48. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 56 τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 61 τροπολογία υπέρ, α, αποσύρθηκε συγγνώμη, 55 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 56 τροπολογία υπέρ, 65 ε, με συγχωρείτε, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αληθεύει αυτό εδώ. 57 δεύτερο τμήμα. 57 λοιπόν. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τοπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τοπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, αποτέλεσμα 27 υπέρ, κανείς εναντίον, καμία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Μιγκάζη. Για να προσθέσω ότι είναι μια από τις σπάνιες στιγμές όπου ο κύριος Μιγκάλσκι ψηφίζει όπως και η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας. <laughs> Ja, wie schon Φτάσαμε στο τέλος των ψηφοφοριών. Περνάμε στο σημείο 9. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που εξεπροσώπησαν άλλους στην ψηφοφορία. Τους ευχαριστούμε και έτσι συνεχίζουμε. I have to go ciao, ciao. Italian boys. Yeah. The Italians said the Italian boys. Not me. Anyway, so Λοιπόν, περνάμε στο 9 τη ημερήσιας διάταξη. Πρόκειται για τον Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό έτος 2013. Έτσι λοιπόν, θα περάσουμε. Ναι, νομίζω καλύτερο να δώσω τον λόγο αμέσω σε εσά, κύριε. Όχι. Ξέρετε όλοι ότι το Συμβούλιο με μεγάλη καθυστέρηση υποβάλλει πάντα τις προτάσεις του. Πιστεύουμε ότι τον Ιούλιο πιστεύαμε θα, ότι θα ερχόντουσαν, τέλη Ιουλίου και τώρα έχουμε τώρα πάλι το πρόβλημα ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν είναι παρόντες επειδή θα έχουμε τις διακοπές, θερινές διακοπές και έτσι θα πρέπει να επιφυλαχθούμε των δικαιωμάτων μας όπως ε, και πέρυσι. Πέρσι είχαμε την εξή διαδικασία που εγκρίναμε. 10 Ιουλίου <clears throat> θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, είχαμε πει, οι τροπολογίες που μπορούν να κατατεθούν μόνο στα αγγλικά θα είναι διαθέσιμες λόγω του ότι είναι πολύ πιεστικές οι προθεσμίες. Πρέπει όμως και από πλευράς Λόκεγκαρντ εισηγητού να δοθεί εντολή. Αν και όταν το Συμβούλιο απορρίψει ή τον προϋπολογισμό μας, τις προτάσεις μας, τις τροπολογίες μας αυτές να τις επανυποβάλει. Και οι, προτάσεις, οι αρχικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής του αρχικού σχεδίου να αποκατασταθούν με αυτή την κατάθεση τροπολογιών. Αυτό τι σημαίνει. Αν έχουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία συμφωνούμε και απορρίπτει το Συμβούλιο και τροποποιεί σημαντικά ή σε σημαντικά τμήματα την τροποποιεί, πρέπει να αποκατασταθεί λοιπόν. Και ο κύριος Λόκεγκαρντ εξ ονόματός μας θα έχει την εντολή να το κάνει αυτό. Αυτό το κάναμε πέρυσι, δεν γίνεται διαφορετικά. Επειδή πάντα με μεγάλη καθυστέρηση υποβάλλει τις προτάσεις του το Συμβούλιο σε σχέση με εμά. Λοιπόν, αν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει κάποιος να την αλλάξει, παρακαλούμε να υπάρξουν τροπολογίες, γι' αυτό στα αγγλικά, εντάξει, και μέχρι τις 28 Ιουνίου πρέπει να έχουν κατατεθεί εδώ. Παρακαλώ να το θυμηθείτε αυτό. Τις χρειαζόμαστε μέχρι τις 28 Ιουνίου. Δεν θα μεταφραστούν στη συνέχεια. Αλλά ας μην περιπλέκουμε τα πράγματα για να μπορούμε όλοι να κατανοούμε τα κείμενα στα αγγλικά και να τα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Έχει τον λόγο τώρα ο κύριο Λόκεγκαρτ. Παρακαλώ κύριε Μόρτεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πλέον τι πρέπει να κάνουμε. Τα περιθώρια είναι στενά. «91 εκατομμύρια ευρώ στο 1α, το έχετε δει αυτό, αλλά βεβαίως ε, στο, στην επικεφαλίδα αυτή υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Αυτό σημαίνει πάντως ότι θα, μοιραστούν τα χρήματα αυτά σε πολλές επιτροπές. Πρέπει να είμαστε σαφές. Η άλλη, επικεφαλίδα είναι το 3β. Εδώ είναι πολύ μικρότερο το ποσό, 25,6, που επίσης θα μοιραστεί και με άλλες επιτροπές. Πάντω είδαμε πέρσι ότι τα περισσότερα από τα χρήματα αυτή τη επικεφαλίδα πήγαν στη δική μα επιτροπή. Μα ενδιαφέρει το 3Β. Εδώ πραγματικά θα πρέπει να βάλουμε σειρά προτεραιοτήτων. Το 2013 είναι το τελευταίο έτος του παρόντος MFF και επομένως ε, για πυρηνικές περιοχές, ε, για πολύ συγκεκριμένε κεντρικές περιοχές έχουμε, ε, πρέπει να τελειώσουμε τις πληρωμές έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σωστά αυτή η προγραμματική περίοδος. Προτείνω λοιπόν αύξηση των δεσμεύσεων και ε, των πληρωμών έτσι ώστε το 2013 να ξεκινήσει το πρόγραμμα κανονικά πέρσι. είχαμε δώσει χρήματα για την διαβίου μάθηση. Ε, εγώ φέτος ε, προτείνω να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στην μείωση. Θα είναι 13 εκατομμύρια ευρώ ε, για το σημείο αυτό. Νομίζω ότι είναι καλή αρχή. Και αν ε, κοιτάξει κανείς και τα δύο προηγούμενα έτη, θα καταλάβει ότι στην ουσία ε, πήραμε αυτό που θέλαμε, άρα οι προϋποθέσεις είναι καλές. Επίσης, αθλητισμός. Ε, σημαντικός ρόλος του αθλητισμού και του σχολικού αθλητισμού ε, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε ε, την χρήση αναβολικών. Έχουμε ήδη κουβεντιάσει, έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα αυτό και νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα να συμφωνήσουμε. Τέλος, επικοινωνία. Μετά από δική μας πρωτοβουλία η Κομισιόν ε, μας ε, ε, δημοσίευσε ένα πολύ ικανοποιητικό έγγραφο στρατηγικής το οποίο αφορά την επικοινωνία. Έχουμε εδώ το πρόβλημα του αποθηματικού βεβαίως. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς είναι οι γραμμές του προπολογισμού, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε ε, να βελτιώσουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας ε, και τις δυνατότητες επικοινωνίας με τους ε, πολίτες. Καλή ευκαιρία λοιπόν να δούμε ποια είναι τα προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται και με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση. Βεβαίως περιμένω και τα σχόλια των ε, μελών και των εισηγητών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λόκεγκάτ. Μάλιστα. Οι συνάδελφοι λοιπόν παρακαλώ να ε, παρέμβουν αν έχουν κάποια παρατήρηση για το πρόγραμμα αυτό. Das ist offensichtlich. Προφανώς. Α, εσύ Σίβο. Εντάξει, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνούμε με όλα όσα ανέφερε ο εισηγητής. Όχι λοιπόν μόνο εσείς συμφωνείτε αλλά και όλοι οι άλλοι επειδή κανείς δεν θέλησε να παρέμβει. Πολύ καλά. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Λόκεγκαρντ όλοι για το έργο που επετέλεσε. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη μάχη που δίνει, για τα μικρά αυτά ισχνά κονδύλια που ζητούμε να μας δώσουν. Η διαδικασία έχει όπως σας περιέγραψα και θα το βρείτε και στους φακέλους σας. Αν δείτε αυτά τα πολλά έγγραφα θα βρείτε τη σελίδα και εκεί υπάρχει το 9. Στο 9 θα βρείτε αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν πότε, α το είπα, στις 12, στις 26, 26 28 διορθώνει η πρόεδρος Ιουνίου, 28 Ιουνίου το μεσημέρι πρέπει να έχουν κατατεθεί τροπολογίες αν επιθυμεί κάποιος να αλλάξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εγγραφό της. Παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ε, μάλιστα, παρίσταται. Κοίταξα αλλού. Εσείς. Ωραίο ότι είσαστε, ότι είσαστε εδώ παρόν. Παρακαλώ. Overall, ε, Ευχαριστώ όλους. Βέβαια, συμφωνούμε συνολικά με αυτά που είπε ο κ. Λουκουβέχτ. Μπορούμε πολύ εύκολα να βολέψουμε αυτά τα επιπρόσθετα ποσά τα οποία ζητούνται για τα προγράμματα διαβιομάθηση. Όντω τα περιθώρια δεν είναι πολύ μεγάλα και όπω ίσως γνωρίζετε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι πληρωμέ, αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα. Ακόμα και για φέτο διακινδυνεύουμε λόγω των ψηφοφοριών των προηγούμενων ετών όπου αυξήσατε τις ε, δεσμεύσεις και το Συμβούλιο περιέκοψε τις πληρωμές. Οπότε τώρα αρχίζουμε και έχουμε πολύ λίγες πιστώσεις και ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα φέτος. Για του χρόνου θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Είναι κάτι λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Συνολικά βέβαια όταν ε, όταν βλέπουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις ή τα πιλωτικά προγράμματα, αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς πραγματικά, θα θέλαμε να ελέγξετε κι εσείς κατά πόσον τα τρέχοντα προγράμματα που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια, μήπως μπορούν ήδη να καλύψουν και τα ε, νέα αυτά προγράμματα, να μην υπάρξει ένας πολλαπλασιασμός πρωτοβουλειών ακόμα που επικαλύπτονται με υφιστάμενα προγράμματα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εάν θέλετε δηλαδή να τονίσετε κάτι ιδιαίτερο σε φυστάμενα προγράμματα, μπορούμε να βρούμε μια μεταφορά πιστώσεων και αναφερθεί συγκεκριμένα στο πρόγραμμα για κάτι. Είναι πολύ καλύτερο αυτό από ότι να υπάρχει πολλαπλασιασμό πολύ μικρών κατακαιρματισμένων πρωτοβουλειών. Και σε ό,τι αφορά βέβαια τη διαχείριση όλων αυτών των έργων, είναι πολύ πιο εύκολο να ενταχθούν σε υφιστάμενα προγράμματα κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτέ τι preparatory actions που έχουν κατατεθεί. Γίνεται προσπάθεια να δούμε τι καλύπτεται, τι όχι. Μπορώ να κατανοήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι πρέπει περισσότερο σε μεγαλύτερα τμήματα να επικεντρωθούμε αλλά ακόμα και τα, οι μικρές πρωτοβουλίες είναι σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν όλα να είναι υπόθεση 200-300 χιλιάδων ευρώ. Πρέπει και σε μικρότερα τμήματα η κονδύλια να μπορούμε κάτι να κάνουμε. Για τους ανθρώπους στις περιφέρειες που με μικρότερες τέτοιες πρωτοβουλίες ε, ε, βρίσκουν κάτι το θετικό δεν πρέπει να περιορίσουμε αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια παρατήρηση που πάντα γίνεται από του συναδέλφους και ήθελα να το πω και εγώ αυτό. Είδα ότι από την DG.com υπάρχει κάποιος παρόν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι κάποιος παρόν. Εσείς είσαστε μάλιστα. Και πάλι θέλω να σας παρακαλέσω αυτό που είπε ο κύριος Λόκεγκαρτ να το διαβιβάσετε στην Επιτροπή, στους ανωτέρους σας. Χαιρόμαστε για το ότι έχει ένα στρατηγικό έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αξίζει αυτού του τίτλου και είμαστε υπέρ σας. Δίνω τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα όσα είπατε βεβαίως θα διαβιβαστούν στο Γενικό μας Διευθυντή. έχω σημειώσει όλα και θα τα διαβιβάσω. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Λοιπόν, ξέρετε όλοι, αν θέλετε να υπάρξει κάποια τροποποίηση, να καταθέσετε τροπολογίες έγκαιρα, όπως είπαμε. Εντάξει, περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι το σημείο 10 και το σημείο 11. Και τα δύο θα καλυφθούν από την κυρία Χρυσούλα Παλιαδέλη. Πρόκειται για το Ίδρυμα Καινοτομία και Τεχνολογία, λοιπόν. Δεν θα σα πω πολλά πράγματα. Δίνω αμέσω τον λόγο στην κυρία συνάδελφό μα, την κυρία Παλιαδέλη. Έχετε τον λόγο, κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, είναι, δύο γνωμοδοτήσεις για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ε, η μία αφορά σε τροποποίηση του κανονισμού του παλαιότερου σχήματος όπως συστάθηκε το 2008. Ε, εδώ οι τροπολογίες ήταν ελάχιστες, ε, αφορούν περισσότερο διατυπώσεις και επικεντρώνονται κυρίως το ρόλο των πανεπιστημίων, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που θα μετάσχουν στην στις λεγόμενες κοινότητες γνώσης και καινοτομίες, τα, τα kicks τα επιλεγόμενα. Έχω μια αγωνία για, το, για την ανεξαρτησία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γενικότερα όταν εντάσσονται σε ομάδες όπου ε, μετέχουν και επιχειρήσεις. Κατανοώ την ανάγκη για την προσαρμογή ορισμένων προγραμμάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις ε, ανάγκες της αγοράς αλλά δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο οι ανάγκες της αγοράς να επιβάλλουν ε, τα δικά τους ετούμενα και να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή ελευθερία των ε, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον κανονισμό ε, και τις τροπολογίες που έχω καταθέσει γύρω στις ε, έξι τροπολογίες για μένα πιο σημαντική είναι ότι για την ώρα η, εκπαίδευση, συνεργασία σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών αυτών των ε, κοινοτήτων γνώσης και καινοτομία θα πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά και μόνο στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Θεωρώ απαράδεκτο να, να υπάρξει προσπάθεια να περάσουν προγράμματα των ε, κοινοτήτων με βάση τα αιτούμενα των, ε, των συμπράξεων αυτών και στην προπτυχιακή εκπαίδευση. Επομένω είναι για μένα πολύ βασικό να περιοριστεί για την ώρα μέχρι ότου εφαρμοστεί η, το πρόγραμμα, τα, να εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά τα κοινά των σπουδών μόνο στην, στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Γιατί από εκεί πέρα προκύπτουν ε, ε δεσμεύσεις για όσους μετέχουν στην, ε, στα προγράμματα αυτά που ίσως ε, υπερβαίνουν τα όρια της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Επομένως, στον κανονισμό δεν έκανα πολλές ε, τροπολογίες παρά μόνο εκείνες που θεωρώ ότι υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία ε, στο μέτρο που μας αφορά. Ε, να πάω στο δεύτερο, κυρία Πρόεδρε, ή να ε, σταματήσω εδώ και να συνεχίσουμε μετά. Που αφορά, το δεύτερο αφορά, η δεύτερη γνωμοδότηση αφορά στη στρατηγική του. Να συνεχίσω. Okay. Το δεύτερο είναι, η δεύτερη γνωμοδότηση αφορά στη στρατηγική ε, στο στρατηγικό θεματολόγιο του, της ε, καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Εδώ ε, ένα μεγάλο κενό που έχει ήδη διαπιστωθεί στην, και σε προηγούμενες συζητήσεις που δυσκολεύομαι βεβαίως να το περάσω με σαφήνεια είναι η απουσία, ίσως γιατί ο όρος καινοτομία και τεχνολογία είναι απαγορευτικός, είναι απαγορευτικός ορισμένων κλάδων της επιστήμης που δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν στις λεγόμενες ε, θετικές επιστήμες. Υπάρχει μία δυναμία στο να συμπράξουν οι επιστήμες των ανθρωπιστικών σπουδών σε αυτού του είδους το θεματολόγιο. Μπορούν βεβαίως να το κάνουν μέσα από την ε, διεπιστημονικότητα και αυτό προβλέπεται. Εκτιμώ ωστόσο ότι και εδώ ακόμη σε αυτό το θεματολόγιο, σε, αυτή τη στρατηγική, σε αυτό το κείμενο, θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για την αναγνώριση των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί ως έναν βαθμό θα επηρεάσει και την, ε, το, θα, ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας ε, στο Horizon 2020, στον ορίζοντα 2020, θα πρέπει η Επιτροπή μας να δώσει ε, και στους συντάκτη, με αυτή την αφορμή του EIT ε, ε, το έναυσμα να ξανασκεφτούν τις ανθρωπιστικές σπουδέ. Έκανα μια ερώτηση με αυτή την αφορμή στην Επιτροπή για τις ανθρωπιστικές σπουδέ και γιατί δεν περιλαμβάνονται με σαφήνεια και στο EIT αλλά κυρίως στον ορίζοντα 2020 και η απάντηση ήταν ότι βεβαίως συμπεριλαμβάνονται. Είναι περίεργο όμως ότι ε, μπερδεύουν στην Επιτροπή και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσουμε το humanities με το humanitarian. Ε, τα humanities είναι κάτι άλλο από το humanitarian. Ε, δεν μπορεί να συμπίπτουν οι ανθρωπιστικές σπουδές με τις σπουδές που ασχολούνται με τον άνθρωπο. Επομένως δεν μπορούν να συμπίπτουν με την ψυχολογία, ή με, την, με το περιβάλλον όπως προέκυψε από την απάντηση που δέχτηκα στην ερώτηση που έκανα στην Επιτροπή. Επομένως, παρόλο που οι ανθρωπιστικές σπουδέ δεν εντάσσονται απολύτως στο σκεπτικό της καινοτομίας, ε, οι τροπολογίες μου ε, έχουν στόχο, θα τις δείτε φαντάζομαι, να φέρουν σε ανάμνηση πάντα την ανάγκη ε, την, για την κατανόησε από τη μεριά της Επιτροπής ότι η έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, επομένως από αυτή την άποψη θα μπορούσε να υποστηριχτεί ακόμη και στο, ε, στο στρατηγικό πλαίσιο του, του Ινστιτούτου. Ε, αν δείτε τις τροπολογίες μου, νομίζω θα καταλάβετε το σκεπτικό μου. Ε, μία ε, τελευταία παρατήρηση ε, αφορά στον ορισμό των νέων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίες για τις επόμενες χρονιές. Πρέπει να γίνει σαφέστερη η διατύπωση, να μας δοθεί ο χρόνος να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το EIT πριν καταλήξουμε για το 2008 ποιες περιοχές, ποιο περι... ποια αντικείμενα επιστημονικά θα προταθούν προκειμένου να δημιουργηθούν αυτές οι, ε, ε, ε σε ποια πεδία θα πρέπει να ε, δημιουργηθούν αυτές οι κοινότητες γνώσης και καινοτομία. Ε, νομίζω ότι τέλειωσε κυρία Πρόεδρε. Αν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις ή ερωτήσεις θα χαρώ πολύ να τις ακούσω. Και περιμένω βεβαίω τις τροπολογίες σας για να εμπλουτιστεί αυτό το δικό μου κείμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Παλιαδέλη. θα έλεγα ένα τροτό σημείο ως αχιλιοπτέρνα τονίζεται που και στα άλλα προγράμματα μας προβληματίζει. Το πρόβλημα το ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες ουσιαστικά κάπως έχουν αμεληθεί, έχουν παραμεληθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 2020 αυτούς ακολουθεί και θέλει να ευδοκιμήσουν και όλα όσα αφορούν την απασχολησιμότητα από πλευράς της δεν ε, συναρτώνται άμεσα με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αμφιβάλλουμε όμως αν αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Γι' αυτό πρέπει να δούμε την δική μας επικέντρωση και εστίαση. Εμείς πρέπει να τονίσουμε να ληφθούν υπόψη αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα τονίσει κανένας άλλος. Εσείς κύριε έχετε τον Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης την εισηγήτρια για τις γνωμοδοτήσει της. Θα ήθελα κάποια σημεία εδώ να τονίσω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και πάλι εκ νέου να τονίσω ότι τον στόχο αυτής τη ε, της Ευρωπαϊκής τον υποστηρίζω για την υλοποίηση δηλαδή του προγράμματος με τον ορίζοντα 2020 να έχουμε ένα σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας που θα μετατεθεί εκεί και παρακαλώ σε σχέση με τα έγγραφα να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι είμαι κατά της περικοπής του προϋπολογισμού των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού ε, Ιδρύματος για Καινοτομία και Τεχνολογία Πιστεύω ότι πρέπει να μπορέσει με πιο ευδιάκριτο χαρακτήρα να ληφθεί υπόψη το ίδρυμα αυτό από τους πολίτες. Αλλά αν περικόψουμε κονδύλια δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε σχέση με τη στρατηγική αυτή της ε, ατζέντα του θεματολογίου αυτού, το υποστηρίζουμε. Παρότι όμως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η ανθρωπιστική πτυχή των ανθρωπιστικών ε, επιστημών. Ε, συμφωνώ με τροπολογίες της εισηγήτριας όπου τονίζει ότι στις ε, περιφέρειες και τα κράτη-μέλη πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες ε, της ε, ε, που να, έχουν, να συμμετάσχουν στις ε, ε, προσπάθειες αυτές όταν δεν καλύπτονται επαρκώ σήμερα. Και για τη συζήτηση στο τέταρτο σημείο η συμμετοχή των νέων κρατών μελών στα ΚΙΚΣ, στις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας δεν επαρκεί και πρέπει να κάνουμε κάτι να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα. Άλλοι θέλουν να παρέμβουν. Κάποιος από την Επιτροπή παρακαλώ. Εσείς. Ποιο από την Επιτροπή εσείς παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Um, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις ε, δύο εκθέσεις αυτές. Έχουμε βέβαια σημειώσει τις προτινόμενες τροπολογίες και νομίζω ότι είμαστε σε επικοδομητικό διάλογο, τον οποίο θα θέλουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καλώς. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Θα έλεγα λοιπόν κυρία Παλιατέλη, κάνατε πολύ καλή δουλειά μετά από τις τελευταίες συζητήσεις κάποιες από τις επιθυμίες μας τις εντάξατε στα κείμενά σας και δεν έχουμε τίποτα άλλο να παρατηρήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα στον ορίζοντα Horizon και μέσω του Ιδρύματος Καινοτομίας και Τεχνολογίας να πετύχουμε τα πανεπιστήμια να δεσμευθούν και να ενταχθούν και αυτά. Εκείνα τα οποία δεν έχουν ακόμα το σύμβολο, το έμβλημα υπεροχής ή αριστείας. Excellence label. Θέλουμε να ληφθεί υπόψη είναι αυτό. Μια συνεργασία μεταξύ εκείνων των πανεπιστημίων που έχουν αυτό το σύμβολο, το έμβλημα Excellence Labor θα πρέπει να οδηγήσει και εκείνοι που δεν συμμετέχουν και δεν το έχουν να μπορέσουν να συνεργαστούν. Σε αυτά τα ιδρύματα και πανεπιστημιακούς φορείς πρέπει να υπάρξει ρόλος πλατφόρμας, ρόλος συνδέσμου για να μπορούν να συνδέουν την πρώτη ομάδα με την δεύτερη. Και στα νέα κράτη-μέλη ή στα υποένταξη κράτη-μέλη υπάρχουν ανάγκε να καλυφθούν τα κενά επειδή είναι πιο χαζοί αυτοί οι εκπρόσωποι αυτών των κρατών μελών, αλλά επειδή δεν είχαν ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα. Να βρεθεί λοιπόν μια τέτοια δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας, να βρεθεί μια τέτοια δυνατότητα για αυτή την πλατφόρμα, για αυτή τη διασύνδεση θα έλεγα με αυτόν τον τρόπο πρέπει να μπορέσει αυτή η άποψη να ληφθεί υπόψη και το θέμα των ανθρωπιστικών ε, επιστημών. Είσαστε στη σωστή πορεία. Ευχαριστούμε την κυρία Παλιαδέλη λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις προθεσμίες ε, πότε θα κατατεθούν στις 28 Ιουνίου και αυτές, μάλιστα, τέλη της επόμενης εβδομάδας. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 28 Ιουνίου. Αν δεν έχετε τροπολογίες δεν χρειάζεται να καταθέσετε τροπολογίες, να μην ε, μακρύνουμε την διαδικασία. Για αυτά τα θέματα όμως θα υπάρξουν κάποιες τροπολογίες από πλευράς μου για να αναφερθεί αυτό το θέμα ρητά και κατηγορηματικά. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σας ευχαριστούμε. Περνάμε στο σημείο 12 Α, ο συνάδελφος Φοντάνα που στην τελευταία συνεδρίαση δεν μπορούσε να παραστεί. Έχουμε το θέμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών. Παρακαλώ, κύριε Λορέντσο Φοντάνα, έχετε τον λόγο. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη φορά κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αλλά η αλήθεια είναι ότι έφτασα πολύ αργά ήταν, και ήταν ήδη και τελευταίο με της ημερησίας διάταξης. Σε βάση περιπτώσει, σα ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτός ο κανονισμός πρέπει να πω ότι είναι ένας ε, καλός κανονισμός, ε, διότι αφορά την διάχυση των διευρωπαϊκών δικτύων ε, τηλεπικοινωνιών. Στόχος του κανονισμού, ο στόχος μάλλον είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, διότι μέχρι το 2020 θέλει να έχει καθολική κάλυψη ε, των, ε, ε, των ευρωζωνικών επικοινωνιών ή 50% των ε, ε, οικογενειών με ε, ταχύτητα σύνδεσης πάνω από 100 MB. Είναι πολύ φιλόδοξο το σχέδιο, αλλά παρόλα αυτά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η τεχνολογική εξέλιξη στην Ευρώπη βεβαίως περνάει μέσα από τις ευρυζωνικές συνδέσεις και συμφωνώ, συμφωνώ με αυτό τον κανονισμό λοιπόν, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Πρέπει να πω επίσης ότι ως Επιτροπή που ασχολούμαστε με θέματα ε, πολιτισμού, αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι ε, να εισάγω σε αυτόν τον κανονισμό την αξία του πολιτισμού μέσα από αυτές τις διασύνδεσεις, γιατί βεβαίως αποτελεί ε, ο πολιτισμός ένα σημαντικό όχημα ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς με τη γνώμοδότησή μας μέσα από τις τροπολογίες μας ε, θα τοποθετηθούμε, ε, θα πούμε δηλαδή ότι μια τέτοια τεχνολογικά εξελιγμένη δυνατότητα επικοινωνίας ε, θα πρέπει να προωθήσει και τον πολιτισμό, να τον ανεβάσει στα μάτια όλων. Να σας πω ότι γενικώ η τροχιά που ακολουθεί αυτός ο κανονισμός με ικανοποιεί γιατί μας κάνει να καταλάβουμε σαφώς ότι εάν θέλουμε να είμαστε σε ίδιο επίπεδο με τον διεθνή ανταγωνισμό, ε, θα πρέπει αν όχι να είμαστε μπροστά από το καιρό μας, τουλάχιστον ε, να ε, ακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών είναι πολύ σημαντικά κατά αυτήν την έννοια. και επομένως από αυτή την άποψη λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να ακολουθεί τα βήματα της τεχνολογικής εξέλιξης για να παραμείνει ε, σε παγκόσμιο επίπεδο σε ανταγωνιστική θέση. Επίσης, ε, ε, ακόμα και στις πιο περιφερειακές, ε, τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, τις ορεινές περιοχές. Και εκεί είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα δίκτυα, να είναι διαθέσιμες αυτού του είδους οι τεχνολογίες, οι οποίες θα διασυνδέσουν τις περιφέρειες αυτές με το υπόλοιπο της Ευρώπης και επομένως οι περιφέρειες αυτές θα μπορέσουν να κρατήσουν τον πληθυσμό τους εκεί. Να μην περιοριστούμε δηλαδή μονάχα στι αστικέ και περιεστικές ε, ε, περιοχέ. Αυτά ήθελα να σα πω τώρα εάν θέλετε να εκφράσετε ιδέε, εάν έχετε κάποια σχόλια, εάν θέλετε να δείτε κάτι οπωσδήποτε στι παρατηρήσει μα, παρακαλώ ε, να μα το πείτε. βεβαίω εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σα, έτσι ώστε να σα ακούσω και να εισάγω στην γνωμοδότησή μου οτιδήποτε μου προτείνετε. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Φερχάν και μετά κυρία Μακλάρκη. Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης έχουμε και πολιτισμικά θέματα και θέματα εκπαίδευσης, παιδείας, κατάρτισης και της διεύρυνσης των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών στα δίκτυα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να πορευθούμε με θετικό τρόπο. Γιατί ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές. Χωρίς επαρκές δίκτυο θα έχουμε μια αποκοπή των ε, περιφερειών και των χώρων της υπαίθρου. Και κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Με εξέπληξε ότι στο σχέδιο ε, έκθεσή σας στην τροπολογία 2 υπάρχει ένα εδάφιο πού να το, πώς να το πω, έχω, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για τις δημόσιες επιχορηγήσεις. Αυτές όμως είναι ακριβώς αναγκαίες, οι επιχορηγήσεις και τα κονδύλια. Εκεί όπου δεν υπάρχουν υποδομές για το δίκτυο ευραίων, ε, το ε, ευρυζωνικό δίκτυο συχνοτήτων, να μην αποκοπούν ε, οι περιοχές της υπαίθρου σε σχέση με τους χώρους των αστικών κέντρων, όπου εκεί υπάρχουν θετικές προσφορές. Πρέπει λοιπόν να πρικοδοτηθούν στον τομέα της υπαίθρου εκεί συνειδητά ο τομέας της εκπαίδευσης παιδείας μέσω του διαδικτύου να μπορέσει να προαχθεί. Δεν γίνεται αυτό σήμερα, δεν υπάρχουν υποδομές αυτές και γι' αυτό στην από την ομάδα μας επιφυλάσσομαι να καταθέσω τροπολογίες για αυτό το στόχο. Με τις προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται ένα σημαντικό ε, βήμα με θέματα που αφορούν αυτά τα θεμελιακά, θεμελιώδου σημασίας ε, θέματα ως προτάσεις, διότι χωρίς τις υποδομές δεν χρειάζεται να κάνουμε λόγο για το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών και του διαδικτύου. Είναι θέμα κοινωνικής σωστής στάθμισης ώστε να προβούμε στην σωστή αντιστάθμιση μέτρων για το χώρο της υπαίθρου και την, ε, τις επαρχίες, τις περιφέρειές μας. Είναι πολύ σημαντικό για το χώρο της υπαίθρου αυτό, τονίζεται και στην έκθεσή σας και είναι σωστό. Χαίρομαι για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτό το θέμα το έχει ενστερνιστεί και το υποστηρίζει και είναι σωστό και αυτό ένα σημείο θέλω να αναφέρω. Την ταχύτητα με την οποία μπορούμε να προβούμε ε, σε κινήσεις στο δίκτυο των 800 ε, ε, κύκλων ευρυζωνικής συχνότητας. Δεν ε, ίσως είναι εύκολο να επιτευχθούν όλα ή έχει δίκιο κύριος Φοντάνα. Είναι πολύ φιλόδοξο αυτό το πλαίσιο να υπάρχει ελεύθερη περιαγωγή, free roaming σε όλες τις ε, περιοχές της Υπέθρου πρέπει να υπάρξει από 30 MB ε, μέχρι το 2020 η δυνατότητα πρικοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συχνότητες αυτές. Έχουμε πολλές τέτοιες περιφέρειες, νησιωτικές περιοχές, τις εσχατιές της Ευρώπης ε, που πρέπει να καλυφθούν. Είναι όμως σωστό να έχουμε φιλόδοξα σχέδια. Πρέπει να δούμε πώς σε συνδυασμό με το δημόσιο, με τον κρατικό τομέα, με τις επιχορηγήσεις και τα κονδύλια που θα διαθέτουν θα πετύχουμε να ε, διαθέσουμε στους πολίτες μας αυτή τη δυνατότητα. Κυρία Μακλάκιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η, Επιτροπή, η προτάση Επιτροπής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, είναι πολύ φιλόδοξες και έχω κάποιο ρολογισμό σε ό,τι αφορά τη διατηθέμενη χρηματοδότηση. Δεν Υπάρχουν πάρα πολλέ πτυχέ πρώτα πρόταση αυτή που μπορούν να μα βοηθήσουν να πετύχουμε του στόχου που έχουμε θέσει για την ψηφιακή ατζέντα μέχρι το 2020. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω την υποστήριξή μου στην έμφαση που δίνεται στο να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να πετύχουν τον στόχο κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο μέχρι το 2020. Είναι απίστευτο στόχος, με δεδομένο ότι κάποιοι δεν έχουν βασική προσφέλαση σε δίκτυα διαδικτύου είναι πολύ αργή η πρόοδο. Ιδιαίτερα στη δική μου περιοχή, τα Ανατολικά Midlands, ε, είναι πάρα πολύ πίσω η όλη κατάσταση. Πρέπει όμω να έχουμε πρόσβαση και στο πλήρε δυναμικό τη ενιαία αγορά. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε πραγματικά αυτή την υποδομή να λειτουργεί για την επόμενη γενιά των τηλεπικοινωνιών. Οι προτάσει που περιλαμβάνουν στον κανονισμό αυτό περιλαμβάνουν και υποστήριξη για το στο πεδίο αυτό. Προβληματίζομαι επίση το ότι ίσως ε, υπάρχει επικάλυψη δαπανών στο πρόγραμμα αυτό. Ίσως πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την ε, διαδικασία, θέλετε, διπλής ε, εφαρμογής για το πεδίο αυτό. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι αν θέλουμε να διαθέσουμε πολύ μεγάλα ποσά χρηματοδότηση για τι τηλεπικοινωνίε και την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, πρέπει να υπάρχει και ισόνομη κατανομή στα κράτη-μέλη στο πεδίο αυτό, ώστε όλοι να μπορέσουν να αυξήσουν τη σχετική ταχύτητα διαδικτύου. Συμφωνώ όμω ότι με τον συγκεκριμένο ότι το διαδικτύο είναι εκπληκτική πλατφόρμα για την προαγωγή της, του πολυπολιτισμικότητα και την εξάπλωση και γνωριμία διαφορετικών πολιτισμών. Και η διασύνδεση με υψηλέ ταχύτητε θα είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για δημόσια κτίρια, πανεπιστήμια, σχολεία κλπ. Έχω κάποιες μικρές προβληματισμούς ό,τι αφορά την τροπολογία 7 που ανέφερα, που αφορά την ε, περιοχή των Uplands και των ε, Midlands. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα αλλάξουμε, ίσως να τους βάλουμε σε περιοχές στόχου 2β και όχι απλώς να ξεχωρίζουμε μια περιοχή. Γιατί πράγμα, πράγμα ε, παραλαμβάνω ενδιαφέρει το θέμα της όνομης κατανομής στα κράτη-μέλη. Σίγουρα μπορούμε να συνεργαστούμε όμω πάνω στο θημείο αυτό με τον κύριο Φοντάνα και του κοιόδης ηγητέ, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση και να έχουμε τη σχετική θετική ανταπόκριση από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ κύριε Φοντάνα. Θα κάνω ίσως μια, μια σειρά από μάλλον αφελείς ερωτήσεις. Η πρώτη, ο κανονισμός αφορά στη διεύρυνση της, ε, της Όσο περισσότερες περιοχές, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, βεβαίως ως Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την, αυτή την πρόταση και αυτή την, αυτό τον κανονισμό. αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, α, πώς να το πω, το δεύτερο στάδιο, η, τη θεματική, ποιος την ορίζει σε αυτή την ε, ευρυζωνικότητα. Είναι κάτι που πάει μαζί στον ίδιο κανονισμό ή προκύπτει στην πορεία. Ε, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα ότι βάλατε την Ευρωπαϊκή ως ε, σημαντικό έτσι, διαδικτυακό τόπο για, ε, για, την, για τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό. Ε, επομένως η ερώτησή μου είναι αυτή. Αν μαζί με την ευρυζωνικότητα προκύπτει και το θεματολόγιο της, ε, ε, των προσβάσεων σε σημεία που μας ενδιαφέρουν εμάς ως Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Yeah, vielen Dank. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον συνάδελφο Φοντάνα πολύ για την πρόταση που υπέβαλε. Πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλη μια φορά δείχνει με σαφήνεια πόσο σημαντικό είναι εμείς να αναμειχθούμε ως Επιτροπή Πολιτισμού σε αυτό το θέμα διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από το θέμα της οικονομικής εκμετάλλευσης του θέματος. Σίγουρα, χωρίς αμφιβολία, σημαντική πτυχή αυτή για τα θέματα υποδομών και ευρυζωνικών ε, επικοινωνιών. Όμως εμείς πρέπει να ενδιαφερθούμε για την κοινωνική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, της ίδιας της κοινωνίας. Και είμαστε ευγνώμονες στον συνάδελφο Φοντάνα για την προσπάθεια επέκτασης των θέματων, των θεμάτων με συγχωρείτε, πολιτισμού και τα πολιτισμικά. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται μόνο για οικονομική εκμετάλλευση και ανάπτυξη, για την διεύρυνση αυτών των δικτύων τηλεπικοινωνιών είναι επίσης το θέμα πώς θα διοργανώσουμε την κοινωνική συμμετοχή των πολιτών με την διαθεσιμότητα τέτοιων δικτύων μέχρι την τελευταία περιφέρεια και εσχατιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική πτυχή αυτή. Έχω κάποιο ερωτηματικό για την τροπολογία 2 και εγώ όπως και με άλλο συνάδελφο, πιστεύω ότι χωρίς δημόσια υποστήριξη, με δημόσια κρατικά κονδύλια και επιχορήγηση, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που θέσαμε ενώπιον μας στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Για να φωνάζουμε και να λέμε όλα αυτά είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν, είναι, δεν επιτρέπεται να γίνει, δεν είναι θετικό. Χωρίς ε, κρατική υποστήριξη θα έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό πιστεύω πρέπει να προσθέσω τη φωνή μου και εγώ σε αυτή την παρατήρηση. Και το άλλο για τις συχνότητες επικοινωνίας πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε με, το δικό μας, ε, με τη δική μας δράση ως ε, Επιτροπής Πολιτισμού πρέπει πολύ αυστηρά να μεριμνήσουμε και να ε, τελούμε σε εγρήγορση και να υποπτεύσουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα θέματα, να καλυφθούν όπως πρέπει και για την επέκταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, να δώσουμε μέγιστη προσοχή σε αυτά. Δεν ωφελούν να συζητούμε μόνο για αυτά τα δίκτυα οικονομικά χωρίς να συζητούμε για το περιεχόμενο αυτών που θα εκπέμπονται μέσω αυτών των ε, δυνατοτήτων. Στο ένα ή άλλο σημείο πρέπει να το τονίσουμε αυτό με τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ συνάδελφος Μάτουλα παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός ανταποκρίνεται σε εκείνα τα οποία εμείς θελήσαμε να πετύχουμε μέσω των στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 με μια ευφυή και αηφόρο ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη. Ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρξει χρηματοδότηση που θα πρέπει να διασφαλιστεί κατά το μέλλον, ώστε οι στόχοι που έχουμε θέσει ενώπιόν μας, η οικουμενική, ας το πω, διάδοση μέσω 30 MB να μπορέσει να επιτευχθεί και είναι κάτι που το καλωσορίζουμε και είναι κάτι το ευκταίο αυτό. Η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών τι αποδεικνύει. Αποδεικνύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτή η στοχοθέτηση σε σχέση με τον ορίζοντα χρόνο, ορίζοντα 2020, μπορεί να είναι κάτι που μπορούμε και να ξεπεράσουμε κιόλα με τις προσπάθειές μας. Γιατί κάνω λόγο για τη χρηματοδότηση. Όταν έχει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στο οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι αναδυόμενες χώρες να ξεπεραστούν από εμάς. Εμείς να τις ξεπεράσουμε και να είμαστε πρωτοπόροι παγκόσμια, προπομπή παγκόσμια. Τότε η ευρυζωνική δυνατότητα και το rapid band θα είναι μεγάλη σημασία για να τα καταφέρουμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, οι τεχνολογίες επικοινωνιών πολλές φορές τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών μας ε, μπορούν να τις καλύψουν και να τις αντιμετωπίσουν. Εκεί όπου οι υποδομές όσον αφορά το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να βοηθήσει, οι υποδομές στο, στην τηλεπικοινωνία μπορούν να βοηθήσουν. Γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε τα θέματα του πολιτισμού, των πολιτισμικών και πολιτιστικών θεμάτων σε αυτόν τον τομέα. Όταν κάνουμε λόγο λοιπόν και βλέπουμε τα πράγματα τεχνολογικά από τις δυνατότητες που μας προσφέρουν, τόσο σημαντικότερο είναι να αναγνωρίσουμε ότι η κατάρτιση και εκπαίδευση είναι αναγκαία και πρέπει να βαίνει εκ με τους ίδιους ρυθμούς με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των τεχνολογιών. Πρέπει να υπάρχει η κατάρτιση για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις υποδομές. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συζήτηση με την Επίτροπο κυρία Νέλη Κρούς που είναι αρμόδια για αυτά τα θέματα και που ευχαρίστω ε, θα έρθει στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για εκείνη. Είναι αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε μια διαδικασία διαβούλευση. Ξανασυζήτησα και είπα αυτά τα οποία ανέφερε εσύ. Αυτή την κατάσταση, αν πέσουμε κάτω από τα 800 megabytes στις συχνότητες και μου το υποσχέθηκε και είπε ότι θα προσέξει ιδιαίτερα αυτό το θέμα διότι αυτές οι συχνότητες και οι παρεμβολές και τα προβλήματα που δημιουργούνται παρεμβολές στις συχνότητες όσον αφορά τις χερσαίες εκπομπές, το θέατρο, το ραδιόφωνο πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια νέα τεχνολογία για να μην υπάρχουν τέτοιες παρεμβολές και όλα αυτά είναι δαπανηρά και πρέπει να μπορέσουν να εξευρεθούν κονδύλια για να πληρωθούν. Μου υποσχέθηκε ότι η ίδια θέτει αυτά τα ερωτήματα και ψάχνει να βρει τις σωστές απαντήσεις. Θέλει να βρεθούν οι απαντήσεις για αυτά τα οποία εμείς φοβόμαστε και οι πολίτες φοβούνται ότι μπορεί να συμβούν. Διότι πολλοί που έρχονται σε επαφή μαζί μας σε σχέση με τη διαδικασία διαβούλευσης θέτουν αυτά τα ερωτήματα και λένε Πώς λέει το Κοινοβούλιο αυτά τα πράγματα και γιατί δεν παραπονούνται οι αρμόδιοι. Υποσχέθηκε λοιπόν να εμπλακεί η ίδια για να βρεθούν λύσεις. Και το θέμα το ευρυζωνικό περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά για πολλούς λόγους και για πολι... λόγους πολιτισμού και για λόγους αποψήλωσης ε, των ε, περιοχών της Υπέθρου και εγκατάλειψης των περιοχών αυτών από τους ε, κατοίκους τους πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και είμαστε σε επαφή με τη γραμματεία το δυνατόν συντομότερα να βρούμε μια ημερομηνία ημερομηνία να προσέλθει εδώ η κυρία Νέλη Κρούς να τα συζητήσουμε. Μετά εσείς κυρία και η Επιτροπή μετά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να προσθέσω κάτι, γιατί όπως ξέρετε είμαι συνεισηγήτρια από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να σας υπενθυμίσω ότι τα διαφορετικά ταμεία είναι ένα έξοχο εργαλείο για να διευρύνουμε την την κάλυψη ε, της εμβέλειας των στόχων αυτών. Αυτός ο στόχος των νέων τεχνολογιών και των δικτύων ε, παρουσιάζονται στα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα των περιφερειών. Στο πεδίο αυτό όμως χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο από ό,τι για άλλες θεματικές. Ακριβώς λοιπόν ε, την επίτευξη αυτού του σκόπου, της επίτευξης ε, πολιτισμού από όλου, πρέπει να επιμείνουμε και ακριβώς από την Επιτροπή Περιφερειών το λέω, να μην το ξεχάσουμε. Πρέπει να διαθέσουμε όλους τους πόρους για να έχουμε ακριβώς να περάσουμε το μήνυμα, για να μπορούμε ακριβώς να έχουμε και πρόσβαση στα διαφορετικά. Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με την τροπολογία 2 που από την Πέτρα και από την Σαμπίνε αναφέρθηκε και εγώ πιστεύω δεν μπορεί να ευσταθεί αυτό την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη Γαλλία έδωσε άδειε κρατικές επιδοτήσεις ε, να δοθούν στην βιομηχανία βίντεο. Αν δίνουμε τέτοιες επιχορηγήσεις στη βιομηχανία των βίντεο, κρατικές επιδοτήσεις και επιτρέπονται αυτές, όμως ε, πολλά περισσότερα θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια για τα θέματα που μας απασχολούν. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και όχι ε, να, να παίρνουμε υπόψη την αντίθετη πλευρά και να έχουμε περικοπές. Είναι σημαντικά τα ευρυζωνικά θέματα για μας και για την κοινωνία και τους πολίτες μας. Πρέπει να δώσουμε συνέχεια λοιπόν. Η Σαμπίνε, μετά η Επιτροπή. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι μικρές κοινότητες έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες να έχουν νομική ασφάλεια όσον αφορά τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες μέσω τέτοιων προγραμμάτων και ενισχύσεων που μπορούν να δοθούν. Υπάρχουν κάποιες ε, κοινότητες που έχουν ε, συνενωθεί στην Ήπεθρο και έτσι κοινωνικά έχουν δημιουργήσει μια ας το πω έτσι εταιρική δομή ώστε να μπορούν να προχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις για τις διαφορετικές τεχνολογίες των δικτύων όσον αφορά τις ε, διάφορες ίνες, ε, διασύνδεση μέσω αυτών των ε, τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων πρέπει να δούμε ότι σε κάποιες ε, δυνατότητες που προσφέρονται αυτό είναι θετικό για τις οπτικές ίνες. Είναι όμως σημαντικό επίσης και οι μικρές κοινότητες να μπορούν να ενταθούν στις υψηλές ταχύτητες και αυτά τα δίκτυα και αυτό δεν γίνεται χωρίς κρατική επιδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Γκρέν από την Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστούμε τον εισηγητή για την παρουσίασή του και για τις διάφορες προτάσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαρίστως να εργαστούμε μαζί του στο μέλλον και βέβαια με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Σημειώνουμε τις διάφορες ε, προτάσεις δεν δει να τίθεται ιδιαίτερα ερωτήματα προς την Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα. Αν επιτρέ... μου επιτρέπετε να διατυπώσω κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση. Θεωρούμε ότι είναι μια οικοδομητική προσέγγιση. Μας αρέσει το γεγονός ότι θέλετε να εξαπλώσετε, ας πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο, τα θέματα, τα πολιτισμικά, σε όλο το κείμενο. Γιατί είναι αλήθεια ότι όταν αρχίσαμε να συντάσσουμε το κείμενο και καθώς προχωρούσαμε, εστιάσαμε ιδιαίτερα πάνω στην οικονομική ανάπτυξη και πιθανότατα να μην λάβαμε επαρκώς υπόψη ε, διατυπώσεις που αφορούν την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Παίρνοντα λοιπόν τροπολογία στην ένα στην σκέψη, που επίση προσθέτει σχετική διατύπωση για τα θέματα πολιτισμού, τι τροπολογίε 5, τροπολογία 5 που είναι στο άρθρο 2, πάλι στο ίδιο πνεύμα, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επικοδομητικέ υποδείξει και συνεισφέρουν σε δική ανάπτυξη του όλου κειμένου. Στην τροπολογία, όπως είπα, δύο, τα σημειώνουμε, σημειώνουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Και προφανώς στην συζήτηση και στο Κοινοβούλιο, τη σημειώνουμε. Στην τροπολογία δύο, για μας είναι, θα θέλαμε ίσως να διατυπωθεί, να διευκρινιστεί στο κείμενο κατανοούμε την πρώτη πρόταση στην τροπολογία 2, που μιλάνε για τις δυνατότητες πρόκλησης ε, στρέβλωση αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Έχουμε μέσα στα παραρτήματα κάποιε τέτοιε παρατηρήσει ό,τι αφορά το ευρυζωνικό δίκτυο. σω δεν είναι κακό να υπενθυμίζουμε στον εισηγητή ότι υπάρχει στην έκθεση. Το δεύτερο κομμάτι όμω τροπολογία είναι κάπω λιγότερο σαφέ. Σω θα πρέπει να επαναξετάσετε τη διατύπωση αυτή για να την διευκρινίσετε ίσως και να την εξαλείψετε και να κρατήσετε μόνο το πρώτο κομμάτι της, ε, την πρώτη φράση. Στην τροπολογία 4 αναφέρεται να αναφέρεται το δίκτυο να ίσως να μην είναι κακό. Στην τροπολογία 6, που είναι ένα κείμενο για το άρθρο 2, που αφορά στις υπηρεσίες, Αναφέρεται ότι επί τη βάση της ε, ε, αηφορίας, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής αηφορίας, μια σειρά υπηρεσιών δεν έχουν αυτή τη διάσταση. Ίσως να περιέζεται λίγο περισσότερο από ό,τι θα επιθυμούσατε σε τέτοιου είδους διατύπωση την εμβέλεια, αλλά βέβαια είναι κάτι που μπορούμε, να σκεφτούμε σε ό,τι αφορά τις απομακρυσμένες ε, περιοχές, upland, έχουμε κάποια θέματα συμπερίληψη του κειμένου και στην ε, πρόταση από την Επιτροπή. Μιλάμε για απομακρυσμένες ε, περιφερειακές περιοχές. Νομίζω ότι εν πολύ καλύπτει αυτού του τύπου τις περιοχές που συζητήσαμε, συμπεριλαμβανομένων και των ορεινών περιοχών. Αλλά και βέβαια και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να επανεξετάσετε. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου από πλευρά τη Επιτροπή, αλλά ευχαρίστω να συνεργαστούμε μαζί σα, να θέσουμε ερωτήματα και είμαστε πάντα στη διάθεση σα να ερχόμαστε να σε επισκεφθούμε όποτε θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Βεβαίως, θα ξαναδούμε την τροπολογία 2, έτσι ώστε να γίνει πιο σαφή και για να δηλώσουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ε, χρειάζονται οι δημόσιες επιδοτήσεις γιατί διαφορετικά οι αν δεν χρειάζονται θα είχαν ήδη την ευρυζωνικότητα και δεν θα, είχα, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Είναι γεγονός επίσης ότι ε, υπήρξε κάποια έτσι ε, σύγχυση όσον αφορά την τάση για, αμοιβαία, για αμοιβαίες επιδοτήσεις. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να έχουμε επικαλύψεις. Οπωσδήποτε λοιπόν ε, θα βελτιώσουμε την διατύπωση. Ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα και Αντιθέτως θέλουμε οι διαδικασίες να είναι απλές έτσι ώστε να είναι και αποτελεσματική, αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Βεβαίως θα λάβω υπόψη μου όλα τα ζητήματα τα οποία ανεφέρθησαν. Βεβαίως ε, θέλουμε να γίνει αναφορά στις ορεινές ε, περιοχές γιατί είναι αυτές οι οποίες αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στο να αποκτήσουν ευρωζωνικό δίκτυο. Αλλά φυσικά όλες ε, οι περιοχές πρέπει να έχουν όλες οι ζώνες της περιφέρειας και οι ε, πολύ απομακρυσμένες περιοχές θα πρέπει να έχουν και αυτές ε, ευρυζωνικότητα. Και για αυτές κυρίως είναι πιο σημαντικός ο κανονισμός αυτός. Τώρα, ε, ποιο θα είναι το θεματολόγιο, τι θα ταξιδέψει στην ευρυζωνικότητα όσον αφορά τον πολιτισμό. Αυτό θα είναι συζήτηση που θα πρέπει να γίνει αργότερα. Αυτό που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι να έχουμε το εργαλείο αυτό έτσι ώστε να γίνουμε τεχνολογικά αλλά και πολιτιστικά ανταγωνιστικοί. Ε, οι κάτοικοι των ε, μειονεκτικών περιοχών εννοώ από άποψη γεωγραφική ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση και να βλέπουν οτιδήποτε βλέπει και οποιασδήποτε άλλος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά μπορούμε να εμπλουτίσουμε και το θεματολόγιο κτλ. Αλλά αυτό αφορά το ίδιο το διαδίκτυο, δεν αφορά το συγκεκριμένο θέμα ειδικά. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκαν και σίγουρα θα με βοηθήσουν στην εργασία μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Λίγη Πρόεδρος. Στις 26 Ιουνίου προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για αυτή την έκθεση, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Παρακαλώ να βιαστείτε αν έχετε κάποιες επιθυμίες για τέτοιες τροπολογίες και αλλαγές. Κλείνουμε το σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη εδώ. Παρακαλώ όλοι όσοι δεν ανήκουν στους συντονιστές να εγκαταλείψουν τώρα την αίθουσα. Θα έχουμε συνάντηση, το συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Διακόπτω για τρία λεπτά, ώστε να εγκαταλείψουν όσοι δεν ανήκουν την αίθουσα.